Αγαπητοί συνάδελφοι, τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίας και τα εγκεκριμένα κείμενα έχουν διατεθεί. Έχετε αντιρρήσεις? Όχι. Wir kommen nun zu den Erklärungen. Είμαστε στις επεξηγήσεις ψήφου. Zur Abstimmung. Σας παρακαλώ. Οι ιδιωτικές συνομιλίες εκτός του ημικυκλίου. kann ε, θέλετε μπορώ να πω και ονόματα έτσι και να σας παρακαλώ ξεχωριστά έναν έναν. Αρχίζουμε. Με την πρόταση μορφή κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της επεξηγής ψήφου. Ο συνάδελφος Μαχ. Παρακαλώ κύριε Μάχα, έχετε το λόγο. Μικρόφων, μικρο, μικρο. Now, yes. Yes. Does it work now? Λειτουργεί τώρα. Κυρίες και κύριοι. δεν μπορούμε να λέμε ότι ο κύριος Γιούνκερ ήταν Πρωθυπουργό σε μια χώρα που ήταν φορολογικός παράδεισος και δεν το γνώριζε. Δεν είναι αυτό όμως το πρόβλημά μου μαζί του. Οι ίδιοι πολίτες της χώρας του πιστεύω ότι θα έπρεπε να διαμαρτυρηθούν να του πούν ότι δεν είναι σωστό κάποιες εταιρείες να έχουν χαμηλότερη φορολογία από άλλες. Αυτό θα ήθελα να συμβεί και στη δική μου τη χώρα, εάν υπήρχε ένα ανάλογο φαινόμενο. Όμως, ο κύριος Γιούνκερ δεν είναι διαφανής. Η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε από εκείνον στο Λουξεμβούργο και τώρα προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι δεν θα θέλει άλλες κυβερνήσεις να κάνουν το ίδιο. Στην πρόταση μορφή ευχαριστούμε. Ο κύριο Ζέλτερ. Δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Dann spricht Frau Η κυρία Γκίλ. Frau uh, Κυρία Γκίλ, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε αμετακίνητοι ως προς την ε, φοροδιαφυγή. Είναι απαράδεκτο μεγάλες εταιρείε να έχουν διευκολύνσεις και να μην ε, συμβάλλουν στον ε, δημόσιο κορβανά, διότι υπάρχει ευνοϊκή νομοθεσία από κάποια κάτι μέλη, επιβαρύνοντας φορολογουμένους. Ο πρόεδρος Γιούνκερ έχει κληθεί να απαντήσει για αυτά και είμαστε βέβαιοι ότι, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Με μια ερευνητική επιτροπή ad hoc μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε όμως καλύτερα τα συμφέροντα των συμπολιτών μας. Γιατί δεν είμαι βέβαιη ότι ήταν το συμφέρον των πολιτών βεβαίως που υποκίνησε τους ε, υπευθύνου για αυτή την πρόταση μορφής ευθύ εξ αρχής. Είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και να είμαστε και διαρκώς στην διεθνή ειδησιογραφία. Γι' αυτό καταψήφισα αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκίλ. Ο συνάδελφος Ποσπισίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταψήφισα την πρόταση αυτή που την βρήκα ακροδεξι... της ακροδεξιάς, την βρήκα λαϊκιστική. Θέλουμε να υπάρχει μια θετική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον και χαίρομαι που μόνο μια μικρή μειοψηφία υποστήριξε αυτή την πρόταση. Ο κύριος Γιούνκερ θα αποδείξει την αξία του επιλύοντα προβλήματα ευρωπαϊκών διαστάσεων, τα προβλήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα της, ε, των φορολογικών παραδείσων δεν είναι θέμα νομοθετικό, είναι θέμα ηθικό και δεντολογικό. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι για τους φορολογικούς παραδείσους, ο τρόπος να το αντιμετωπίσουμε αυτό δεν είναι με περισσότερο διοικητικό άχθος, αλλά με ανακούφιση του φορολογικού βάρους ε, για όλους τους πολίτες της Ευρώπης και κρατώντας βεβαίως εδώ τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες. Μην τους δίνουμε κίνητρα να φύγουν και να αναζητούν φορολογικούς παραδείσους. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μορβάη τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως δικηγόρος Σκεφτόμουν ότι αν κάποιος πάει να διαπράξει κλοπή ή διάρρηξη και τον πιάσουνε, τι θα πει, θα αρχίσει να εξηγεί ότι η νομοθεσία δεν είναι καλή και ότι δεν υπήρχαν οι σωστοί νόμοι. Εάν κάποιος ε, σφετεριστεί την ιδεκτουσία άλλων, την αρπάξει, ε, υπάρχει αρπαγή και υπεξαίρεση. Δεν μπορεί να λέει όμως κανείς ότι ο ορισμός στον νόμο δεν είναι σωστός εάν είναι ειδικό και εμπειρογνώμων επί των κλοπών και των διαρρήξεων πώς γίνεται μετά να είναι μέλος ενός σώματος που υψώνει τη φωνή του κατά της κλοπής κατά της υπεξαίρεσης. Υποστήριξα λοιπόν αυτή την πρόταση μορφής και Νομίζω ότι ο κύριος Γιούνκερ δεν είναι ο κατάλληλος για αυτή τη θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Μόρβαη. Ο συνάδελφος Μπάλτσο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, είχαμε την πρόταση Μομφής η οποία απορρίφθηκε Κάτι που αποτελεί ντροπή για μας εδώ. Ο κύριος Ιούνκερ είναι ένοχος διότι κατά τη θητεία του ως Πρωθυπουργό το Δουκάτο του Λουξεμβούργου έγινε φορολογικός παράδεισος και έτσι στέρισε εκατομμύρια ευρώ από ανθρώπους στις χώρες στις οποίες ε, λειτουργούν αυτές οι εταιρείες. Αυτό είναι ντροπή και είναι ντροπή η πλειοψηφία αυτή ε, διότι τα επιχειρήματα υπέρ του κυρίου Γιούνκερ δεν ήταν επιστικά. Έγιναν επιθέσεις σε αυτούς που υπέβαλαν αυτή την πρόταση μομφής. Ε, θεώρησαν ότι θα ήταν πολύ κακό εάν θα έπρεπε να δημιουργηθεί τώρα νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζω όμως ότι είναι αξιόπιστοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι θεματοφύλακα ε, ε, ε, της συνθήκης, σε υποθεσεις τις συνθήκες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Ιγκλέσιας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα δεν είδαμε κάτι καλό σήμερα. Μια πρόταση μορφή στο Κοινοβούλιο την κατέθεσαν αυτοί που είναι υπέρ των φορολογικών παραδείσων, τη City του Λονδίνου δηλαδή, που είναι κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είδαμε και κάτι πιο θλιβερό. Οι σοσιαλιστέ εδώ μέσα και ιδιαίτερα οι Ισπανοί σοσιαλιστέ είχαν την ευκαιρία να υποστηρίξουν την πρόταση μορφή που θέλαμε εμεί να προωθήσουμε κατά τη δυνατότητα ε, των φορολογικών παραδείσων και κατά του υπετίου ε, αυτών των πολιτικών που ε, ζημίωσαν του ευρωπαϊκού λαού. Ξανά έδειξαν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές ότι έχουν μεγάλο ε, πρόβλημα και δυσκολία να περάσουν από τα λόγια στα έργα. Αυτή την εβδομάδα απέδειξαν ότι είναι στο πλευρό του Γιούνκερ και των φορολογικών παραδείσων. Αυτό είναι κακή είδηση για τη δημοκρατία και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Ιγκλέσιας. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, οι ευρωσκεπτικιστέ και η ακροδεξιά υπέβαλαν αυτή την πρόταση μορφή κατά του κ. Γιούγκερ, αλλά με την ίδια ακριβώ συλλογιστική που υποτίθεται ότι θέλουν να καταπολεμήσουν. Δηλαδή, να ε, ε, βάλουν πρώτους τους εθνικούς ε, εγωισμούς και τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών πριν από το ευρωπαϊκό συμφέρον. Ναι, ο κύριος Γιούνκερ πήρε μέρος σε ένα σύστημα που ήταν σκανδαλώδες διότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν φορολογική παράδοση με την ε, χρήση κάποιων εσόδων που δεν φορολογούνται για να τα εκμεταλλευτούν χρηματοπιστωτικοί όμιλοι ή ε, πολυεθνικές εταιρείε. Με τα προγράμματα λιτότητας, με την μείωση των εισοδημάτων στις ε, πιο αδύναμες χώρες, με την διαφυγή ε, εσόδων. Αυτό ε, είναι πολύ ε, εύκολο να το επιρρύπτουμε ένα στον άλλον. Σίγουρα πρέπει να υπάρξουν τιμωρίες. Σίγουρα το σύστημα του Λουξεμβούργου ή αλλού μπορεί να είναι νομοφανές, αλλά είναι ένα σύστημα παράνομο και δεν μπορούμε να διαφύγουμε από τέτοια προβλήματα μόνο αν, παρά μόνο αν υπάρξει περισσότερη Ευρώπη και καταπολέμηση αυτών των φαινομένων προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ, συνάδελφε Ντουιρό. Ο συνάδελφος Χάναν. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Καταψήφισα ε, την, τον διορισμό του κύριου Γιούγκερ, καταψήφισα και την Ευρωπαϊκή του Επιτροπή. Ε, νομίζω ότι ε, να μόνο ειλικρινής ε, στην καταψήφιση του, διότι είναι ένα απομεινάρι από το 1950 που μιλούσαμε για εναρμόνιση ελάχιστων μισθών κλπ. Παρόλα αυτά, όπως σε κάθε άλλος, έχει ε, δικαίωμα στο τεκμήριο αθωότητας ε, και έχει ξεκινήσει η έρευνα και δεν έχει ολοκληρωθεί. Ε, είναι λοιπόν κακή η χρονική στιγμή αυτής της πρότασης Μόμφης και κακή η σύνταξή της επίσης. Δεν μπόρεσα να την υποστηρίξω παρά όλους τους λόγους που έχω να θέλω να ξεφορτωθώ τον κύριο Γιούγκερ εκτός εάν αποδειχθεί ότι έχει κάνει κάτι παράνομο. Ε, οι συνάδελφοι ε, το έχουν παραξηγήσει αυτό. Δεν είναι ε, έγκλημα το να μειώσει κανείς τη φορολογία και εάν κανείς θεωρεί ότι είναι πρόβλημα ότι κάποια άλλη χώρα έχει χαμηλότερη φορολογία μπορεί να μειώσει τους δικούς του φόρους. Ευχαριστώ συνάδελφε Χάνων. Ο κύριος Μαριά, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ως γνωστόν έχω καταψηφίσει τον Γιούνκερ υποψήφιο πρόεδρο της Επιτροπής γιατί ως εκπρόσωπος του παλιού πολιτικού κόσμου της ευρώπης και επί χρόνια πρόεδρος του eurogroup είναι υπεύθυνος για τα μνημόνια την ανθρωπιστική κρίση στην ελλάδα και το επονίδιστο χρέος που φορτώθηκε στις πλάτες του ελληνικού λαού. η αποκάλυψη του juncker gate καθιστά πλέον διπλά επιβεβλημένη την απομάκρυνση του κυρίου juncker. υπερψήφισα λοιπόν την πρόταση μορφής κατά της επιτροπής που υπέβαλε ο κ. zanni και το κίνημα των πέντε αστέρων προκειμένου να απαλλαγούμε από τον juncker και την παρέα του το γεγονό ότι η πρόταση μορφή υπογράφτηκε και από βουλευτέ τη άκρα δεξιά, με του οποίου, ω γνωστόν είμαστε απέναντι και μα χωρίζει άβυσο σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο δεν μπορεί να αποτελέσει άλοθη προκειμένου να μην υπερψηφιστεί η πρόταση μορφή μια και το μείζον διακύβευμα είναι η αποπομπή του juncker. άλλωστε η πολιτική διαδρομή του καθενός είναι γνωστή και καταγεγραμμένη και ω εκ τούτου δεν χωρούν παρερμηνίες όλα τα άλλα είναι υπεκφυγές και εδραιώνουν τον juncker στην προεδρία της επιτροπής. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαριά. Ο κύριος Γιάρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφρίκτού και αρχίζει με την παρακολούθηση της πραγματικότητας και αν δεν μου αρέσει η πραγματικότητα θα την αλλάξουμε με την πολιτική μας ε, της νομοθεσίας. Ε, δεν μας αρέσει η φορολογική πολιτική αυτό το καιρό, συμφωνούμε όλοι, αλλά θα πρέπει να την αλλάξουμε, να την εναρμονίσουμε. Γι' αυτό επιθυμώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάρα πολύ γρήγορα, λυτή δηλαδή, να εργαστεί από αυτού του προβλήματος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παραμείνει ε, λειτουργική. Γι' αυτό καταψήφισα την πρόταση μορφή. Κατά τα άλλα, περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον να δω τι κάνουν τώρα τα κράτη-μέλη. Τι στάση θα τηρήσουν και ε, ελπίζω να χρησιμοποιήσουν αυτή τη φόρα που έχει πάρει τώρα η Ευρώπη για την εναρμόνιση της φορολογικής πολιτικής και να ε, κόψουν τις αντιστάσεις τους στα κράτη-μέλη. Εκεί θα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει και να παραμείνει η λειτουργική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό δεν βοηθάει, ούτε είναι κάτι που μπορεί να τελεσφορήσει μια τέτοια πρόταση μορφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φων Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ υπερψήφισα την πρόταση Μομφής και καταψήφισα τον κύριο Γιούνκερ και την Επιτροπή του. Εγώ θα ήθελα ε, να συνεχιστεί ε, ανεξάρτητα η έρευνα των κατηγοριών αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό δεν συμφέρει την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου που ε, δεν θέλει να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα. Το θέμα είναι νυφάλαιο ε, δεν είναι ιδεολογικά φορτισμένο, δεν είναι θέμα δεξιά ή αριστερά. Υποστηρίζουμε αυτή την επιτροπή ή όχι. Είναι αντικειμενικά τα πράγματα. Εμεί από την εναλλακτική για τη Γερμανία ήδη δύο φορές ε, καταψηφίσαμε ρητά και τον κύριο Γιούγκερ ω πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και καταψηφίσαμε το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό είναι συνεπές ε, και χωρί καμιά ιδεολογική φόρτιση το γεγονό ότι καταψηφίσαμε και πάλι. Είμαστε λοιπόν υπέρ τη πρόταση μορφή και δεν είναι δεξιά-αριστερά τα πράγματα, είναι ε, νυφάλια και αντικειμενικά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φωνστόρχ, ο κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα καταψήφισα την Επιτροπή Juncker Καταψήφισα την Επιτροπή Γιούνκερ για όλους τους λόγους που αναφέρει και η πρόταση μορφής και πρόταση την οποία συνυπέγραψα με τους εκπροσώπους του κινηματός μας και με άλλους συναδέλφους. Επειδή έχω άμεση γνώση των θεμάτων αυτών από την Επιτροπή Περιβάλλοντο αυτό το κοινοβουλίο και επειδή είμαι συντονιστή για τα θέματα αυτά από το κόμμα την ε, Δημοκρατία της ε, την Ευρώπη για τη Δημοκρατία και την Ελευθερία. Ε, και επειδή συζητούμε όλα αυτά τα συστήματα, βλέπουμε ότι οι επίτροποι που έχουν προταθεί δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα ορεκτά κάψιμα και την εξάρτησή μα από αυτά. Στην Ιταλία όμω θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτηση τη χώρα από το πετρέλαιο και βεβαίω τι λαβερέ συνέπειε για τη ζωή των πολιτών. Όπω επίση δεν υπάρχει καμία πρόθεση να μειωθούν οι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου από τι επιχειρήσει τη ΕΕ. Η Επιτροπή του Juncker θέλει επίση να ισοπεδώσει τι ελάχιστε αισιόδοξε ελπιδοφόρε νομοθετικέ προτάσει όπω για τη μείωση του διοξιδίου Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ συνάδελφε Πεντετσίνη. Ο κύριος Κόρνης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψήφισα την πρόταση μου ε, του Πρόεδρου Γιούνκερ και ψήφισα υπέρ όχι μόνο ε, από προσωπική έχθρα εναντίον του σε καμία περίπτωση, αλλά για όλου του λόγου καχυποψία εναντίον του. Να δώσω μερικά παραδείγματα από τα ίδια του τα λόγια. Τα λόγια του κυρίου Γιούνκερ. Όταν μιλήσαμε για τη φοροδιαφυγή και όταν μιλήσαμε για την περίπτωση του Λουξεμβούργου, το θύμισα τότε ότι ήταν ο Υπουργό Οικονομία τη χώρα αυτή και ότι υπήρχαν σκάνδαλα των ε, Λουξεμβουργιανών υπηρεσιών ε, και ότι τότε είχε αναγκαστεί να παρέτηθει και, το, και επισήμανε όλα αυτά τα θέματα. Να πω ότι μου απήντησε ότι ουδέποτε ήμουν υπουργό οικονομία και ουδέποτε παρετήθη. Μα θα έπρεπε, λέει ότι θα έπρεπε να είστε περισσότερο. Μου είχε πει θα έπρεπε να είστε ενημερωμένο και να προσέχετε τι λέτε. Ήταν υπουργό ε, οικονομικών ε, εργασία και απασχόληση. Ήταν 18 χρόνια πρώτοπουργό. Και μετά την παρέτησή του ουσιαστικά οδηγήθηκε σε πρόορες εκλογές. Και βεβαίως ο... φαντάζομαι ότι παρόλο που ο διαδοχός του ήταν στη θέση του, ο ίδιος θα έπρεπε να έχει υποβάλει την παρέτησή του στο Μεγάλο Δούκα. Ευχαριστούμε κύριο Γκόλμης. Ολοκληρώσαμε έτσι τις επεξηγήσεις ψήφου για ε, την πρόταση μομφής ε, κατά της Επιτροπής ε, και τώρα έχουμε επεξηγήσεις ψήφου σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 και δίνω το λόγο στη συνάδελφο Τζιλ. Γκίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό διότι οι καθυστερήσει στην εκκίνηση τη πολιτική συνοχή σημαίνουν ότι στην Αγγλία μπορεί να μην εγκριθούν τα σχετικά προγράμματα. Και ένα από του βασικού λόγου είναι ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει παράσχει τα μέσα για την ε, εκτέλεση των ε, ταμείων. Ε, και αυτό σημαίνει ότι το, η κυβέρνηση Ε, διακυβεύει 900 ε, εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, στην περιοχή μου για την ανάπτυξη των πόλεων μας. Των πόλεων μας. Φαίνεται ότι το βασικό εμπόδιο είναι ο δισταγμός της κυβέρνησης να αναθέσει σε άλλους αρμοδιότητες σχετικά με το πρόγραμμα αυτό που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Γκίλ. Έχετε επεξηγήσει ψήφου για όλα τα επόμενα θέματα και είσαστε η πρώτη ομιλήτρια. Παρακαλώ να είστε έτοιμοι. Ο συνάδελφος Στεχόφσκι. Πρόεδρε, συνάδελφοι, υπερψήφισα την πρόταση αυτή διότι πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε ε, τον μέγιστο αριθμό επιχειρησιακών προγραμμάτων ώστε να επιταχυνθεί η εφαρμογή τους, διότι ήδη έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να διατεθεί επιπλέον χρηματοδότηση ακόμα και το 2015. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Σας θαυμάζω για τον, λόγο που, για τον τρόπο που προεδρεύετε σε αυτή τη συνεδρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν υπέρ της πρότασης αυτής, διότι η πολιτική συνοχής είναι πολύ σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό στήριξα αυτήν την πρόταση και είναι απολύτως ε, ευθυγραμμισμένη με την ε, πολιτική και το πακέτο του ε, Προέδρου της Επιτροπής Γιούνκερ. Ιδιαίτερα σημαντική για μένα είναι η συνεργασία με την Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ο συνάδελφος Στεχόφσκι ήδη αναφέρθηκε στην καθυστέρηση για το διάστημα 2014-2020 και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος και για τους δικαιούχους, διότι τα κράτη-μέλη μπορούν έτσι να αναθεωρήσουν τις ε, συνεισφορές τους. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Πόλτσακ, ε, ο συνάδελφος Ποσπισίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ψήφισα υπέρ από του ψηφίσματος και το συνυπέγραψα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό ψήφισμα, διότι όπως υπόθηκε, αυτή τη στιγμή Έχουμε πρόβλημα με, τις επιμέρους, ε, με τα επιμέρους προγράμματα των πολιτικών συνοχής, ιδίω για το διάστημα του 2014. Το θέμα του Ταμείου Συνοχής και των κονδυλίων της είναι πολύ σημαντικό, ιδίω για τα οικονομικώς αδυναμότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κονδύλια αυτά είναι σημαντικά ε, ως προς τις επενδύσεις και την ροή κονδυλίων για τις υποδομές. Ε, έρχομαι από τη Δημοκρατία της Τσεχίας και μπορώ να σας δώσω κάποιους αριθμού για τη χώρα μας από την προσχώρησή της, λόγου χάρη το δικό μας κράτος κέρδισε περισσότερα από 343 δις κορώνες πέραν του, ε, της συνεισφοράς μας προς τον ευρωπαϊκό προπολογισμό από ε, το πλεόνασμα. Αυτά τα κονδύλια ε, τελικά ήταν ωφέλιμα για τις δικαιωτικές χώρες παρά τα κάποια προβλήματα απορρόφησης. Γι' αυτό πρέπει πάντα να τα αξιοποιούμε. Ευχαριστώ και τώρα κυρία Κίρτον Τάλινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ υπερψήφισα το, ψήφισμα αυτό γιατί είμαι από την βόρειο-ανατολική Αγγλία που λαμβάνει χρηματοδότηση εκατομμυρίων στερλινών και υποστηρίζονται έργα από τα κοινοτικά κονδύλια. Ε, έχουν δημιουργήσει θέσει εργασία και συνεχίζουν να το πράττουν. Βοηθούν την οικονομία και τι δεξιότητε. Και η καθυστέρηση των πληρωμών του Ηνωμένου Βασιλείου διακινδυνεύει τη συνέχιση αυτών των προγραμμάτων και δεν μπορεί μονομερός να καταργήσει ε, τις, ε, τους περιφερειακούς οργανισμούς και όχι μόνο να έπραξε αυτό αλλά ε, επιπλέον ε, καταστρέφει την περιφερειακή πολιτική και η δική μου εκλογική περιφέρεια είναι ακριβώς στο κέντρο ε, αυτής της δίνης. Καλό τις ε, κυβερνήσεις να δείξουν ευθύνη και να λυθεί το συντομότερο δυνατό το πρόβλημα. Έχουμε την υψηλότερη ανεργία και ανεργία των νέων στη Ηνωμένο Βασίλειο 724 ε, ε, εκατομμύρια στελίες διακυβεύονται το επόμενο διάστημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπέρτερ. Ευχαριστώ, η συνάδελφος Μπέρτερ. Ε, στηρίζω την ε, πρόταση μομφή όσον αφορά την καθυστέρηση τη εκκίνηση τη πολιτική συνοχή. Θέλω να στείλω ένα σαφέ μήνυμα προ την Επιτροπή και προ τι κυβερνήσει. 400 ε, εκατομμύρια λίρες ε, στην Αγγλία διακυβεύονται που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, για να καταρτήσουν νέους ανθρώπους, να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και να δημιουργήσουν υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να επιταχύνει τη διαδικασία αυτή και να επιτρέψει να ξεκινήσουν στην ώρα τους τα προγράμματα αυτά. Θα πρέπει να ακολουθούμε τις διαδικασίες, θα πρέπει όμως να υπάρχει κάποια ευελιξία. Θα πρέπει να φροντίσει να ξεκινήσει η εφαρμογή όσο αμέσω μόλι συμφωνήσουν επί της αρχής πάνω στα προγράμματα έτσι ώστε οι τοπικές αρχές να μπορούν να ξεκινήσουν τα προγράμματα αυτά όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ κυρία Μπέρτερ. Ο συνάδελφος Χάνεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, τα προγράμματα της συνοχής θα πρέπει να θεωρούνται από τα πλέον μετρήσιμα και συγκρίσιμα, διότι αυτό το ορίζει και η συνθήκη του Μάστριχτ. Ε, μεταξύ των 11 ε, πλέον αδύναμων περιοχών υπήρξε και μεγαλύτερη ροή κονδυλίων. Ποιο ήταν ο μεγαλύτερο δικαιούχο Ευρωπαϊκών Κεφαλαίων, βεβαίω, η Ελλάδα. Και τι αποτέλεσμα έδινε αυτό. Εάν φορολογούμε τι πλουσιότερε χώρε για να πληρώνουμε τι φτωχέ, τελικά έχουμε λιγότερε πλούσιε χώρε και περισσότερε φτωχέ. Ε, τα κράτη, όταν είναι φτωχότερα μπορεί τελικά να γίνουν εξαρτημένα από τι επιδοτήσει και τελικά δεν εξηγαίνουν τα δικά του δημοσιονομικά επειδή μαθαίνουν να λαμβάνουν δωρεέ. Ακούσαμε από Βρετανού συναδέλφου πόσο σημαντικό είναι να παίρνει κανεί ε, κονδύλια για προγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμω δεν είμαστε απλώ από του ε, βασικού συνεισφέροντε από το Ηνωμένο Βασίλειο ε, και δεν μπορούμε να μετράμε μόνο τα ωφέλη, αλλά και τους, θα πρέπει να μετράμε και τους φόρους. Ούτε μπορούμε να διαφημίζουμε έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να κοιτάζουμε να τονώσουμε την ε, τοπική ανάπτυξη. Εάν θέλαμε να υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρώπη, θα έπρεπε να προάγουμε την ε, διαφορετικότητα, την ποικιλία και την πολυφωνία. Να αφήσουμε τι ευρωπαϊκέ χώρε να ξανάρθουν στι αγορέ μόνε του και να εξάγουν από αυτέ. Και όχι να στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Χάναν, ο κύριο Γιάρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισμα το ψήφισμα θέλω να κάνω μερικέ παρατηρήσει. Πρώτον, η πολιτική συνοχή είναι σημαντική και βοηθάει ε, να συγκλίνουν οι συνθήκες διαβίωσης. Βέβαια, το better spending σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων. Στη δική μου περιφέρεια η πολιτική συνοχή όχι μόνο έχει πιάσει τόπο, αλλά έχει κινητοποιήσει και εξελίξεις. Στην Ανατολική Γερμανία τα νέα ε, κράτη σιγά σιγά βγαίνουν από τον στόχο 1 ε, και ε, αυτό είναι και χάρη στην Ευρωπαϊκή Πολιτική συνοχή. Είναι γεγονός ότι κάθε 7 χρόνια βλέπουμε τα ίδια πράγματα ε, και θα πρέπει πολιτικά να αποφασίζονται μεταβατικές περίοδοι για να μην βλέπουμε αυτή την εμπλοκή και τη στενοπό. Και παρακαλώ τα κράτη-μέλη επιτέλους να δώσουν τις συνεισφορές τους που καθυστερούν τις πληρωμές για να έχουμε τα χρήματα για αυτή την εξαιρετικά επιτυχή πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Γιά. Εδώ τελειώσαμε τις επεξηγήσεις ψήφου για την πολιτική συνοχή 2014-2020 και ερχόμαστε στις κατευθυντήριες Μάλλον, συγγνώμη, στην 25η επέτειο της Σύμβασης του ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. κυρία Αγγίλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ε, με όλη μου την καρδιά στήριξα αυτή την πρόταση ψηφίσματο, διότι συμφωνώ απολύτω στα δικαιώματα των παιδιών. Θα έπρεπε να βρίσκονται στον πυρήνα τη κάθε πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα απέσια νέα για την παιδική κακοποίηση, εκμετάλλευση και παραμέληση, αδιαφορία, ε, δείχνουν ότι υπάρχει κατ' ανάγκη να λάβουμε επιπλέον μέτρα για να προστατεύσουμε τα παιδιά μα. Όλα τα παιδιά, όπου και αν βρίσκονται, ε, όποια κοινωνική και εθνοτική προέλευση και αν έχουν, θα πρέπει να έχουν το ύψιστο επίπεδο μόρφωσης και φροντίδα. Και πιο συγκεκριμένα η προστασία των ανηλίκων είναι κάτι που πρέπει να ε, ενταθεί, διότι είναι από τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που υποφέρουν από, τις, από τους ανεπαρκείς μεταναστευτικούς νόμους και πολλές φορές πέφτουν θύματα των κενών των πολιτικών μας που δεν είναι αυτές που πρέπει. Ευχαριστούμε ο συνάδελφος Κάρφη. Ευχαριστώ. Στήριξα το ψήφισμα για την 25η ε, επέτειο της Σύμβασης του ΙΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και καλωσορίζω την ευκαιρία να σκεφτούμε ότι θα πρέπει σε πρώτη θέση στις προτεραιότητές μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι τα δικαιώματα των παιδιών. Θα πρέπει αυτά τα δικαιώματα διεθνώς να φροντίζουμε να προστατεύονται ώστε όλα τα παιδιά να έχουν δικαίωμα να ζουν και να έχουν μια παιδική ηλικία πέρα από πολέμους ή από άλλε φρικαλαιότητε που μπορεί να γνωρίσουν. Θα πρέπει να υπάρξει μια νέα προσοχή για τα θέματα των παιδιών, μέρημνα για τους νέους, διότι αυτοί πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα για την κρίση και τις ε, ανελαίτες πολιτικές λιτότητας. Σας ευχαριστώ. Αυτός είσαι. Ευχαριστώ κύριε Κάρθη. Ο συνάδελφος Μοργάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα, με την αφορμή της 25η Εμπετίου της Σύμβασης του για τα δικαιώματα του παιδιού, επανέλαβε με ένταση την απόλυτη ανάγκη να προστατευτούν τα παιδιά και να φροντίσουμε πολιτικές της Ένωσης να εγγυώνται την προστασία και την ευημερία των παιδιών. Είναι μια επανάληψη αυτό, αλλά δεν ήταν μια τελετουργική επιλογή. Ε, θα πρέπει να δούμε ποια είναι πραγματικά η κατάσταση στη συγκεκριμένη περίπτωση και πώς το κείμενο που εγκρίθηκε δεσμεύει για στόχους για τα δικαιώματα των ανηλίκων. Ιδίως 25 χρόνια μετά την εφαρμογή της σύμβασης αυτή να δούμε και τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά αποτελέσματα με συγκεκριμένους δείκτες και επίσης να δούμε από όσα είχαν εκφραστεί εκεί κάποια πράγματα λάβαν σάρκα και οστά τι αλλαγή υπήρχε στην οτροπία, στις υπηρεσίες, στην οτροπία και στην, ε, στο εκπαιδευτικό σύστημα για την προστασία των παιδιών και τις οικογένειές τους. Το να μιλάμε για δικαιώματα ανηλίκων και για παιδιά είναι σημαντικό για το μέλλον της κοινωνίας μας. Πρέπει να φροντίσουμε το κείμενο του ψηφίσματος που ψηφίστηκε. κύριε Μπονκάνο. Κύριε Πρόεδρε, Γιορτάζουμε την 25η επέτειο της ε, σύμβασης ε, του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και καταδικάζω τα αποτρόπια πράγματα που συμβαίνουν ε, σε όλο τον κόσμο. Έχουμε υποσυτισμό των παιδιών, έχουμε παιδιά στρατιώτες, παιδιά σε αποστολές αυτοκτονίας και ακούσαμε τα, τα, τις πρόσφατες αποτρόπες πράξεις της Μπόκο Χαράμ στην Ιγυρία, στο Ιράκ ε, τους βιασμούς ε, που γίνονται. Υπάρχουν όμως κάποιες πτυχές ε, του ψηφίσματος που με ανησυχούν. Τα κράτη-μέλη και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη βασική αρμοδιότητα εδώ πέρα και εγώ είμαι πατέρας τριών μικρών παιδιών και πιστεύω ότι κάποιο από τα θέματα που έχουν να κάνουν με την φιλετική ιδιότητα των παιδιών είναι θέμα των ε, γονέων, γι' αυτό, ε, γι αυτό απήχα. Ευχαριστώ, συνάδελφο Γιάρ. Κύριε Πρόεδρε, ε, θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Καταρχάς, η παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού είναι πρόβλημα όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι κάτι που βλέπουμε και σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, στην Επιτροπή Αναφορών, όταν Μιλάμε για τα δικαιώματα του παιδιού. Τα κράτη-μέλη πάντα ε, παραπέμπουν ε, στην ε, δική τους αρμοδιότητα και τρίτον, όσον αφορά τα δικαιώματα του παιδιού, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εισάγουμε μια πιο γρήγορη διαδικασία, διότι ε, το δικαίωμα είναι ένα πράγμα, αλλά ε, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων αυτών είναι άλλο θέμα και ε, δεν είναι καλό για τα παιδιά αν αυτές οι διαδικασίες διαρκούν πολύ χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν πάνω σε αυτό να εργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε Γιάρ, ο συνάδελφος Κέλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα δικαιώματα των παιδιών, ιδίως ένα τόσο σημαντικό έτος, 25 χρόνια μετά την έγκριση και την κύρωση της Σύμβασης του ΙΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Βεβαίω πρόοδο έχει γίνει σε, πολλά, σε πολλές περιοχές, αλλά πρέπει να γίνουν κι άλλα. Ιδίω ό,τι αφορά την εκπαίδευση, το σύστημα υγεία και την ισότητα των παιδιών. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, θα πρέπει πρόσβαση να έχει το κάθε παιδί στο εκπαιδευτικό σύστημα και αργότερα και στην αγορά εργασία. Αλλά και για την υγεία το ίδιο ισχύει. Χωρί υγεία δεν μπορεί κανεί να έχει μια ευτυχισμένη ζωή. Και βεβαίω και για την ισότητα. Η ισότητα των φύλων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου δεν είναι κατεγγυημένο, όπω είπε ο κ. Τάνοκ μόλι τώρα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, κάνουμε κάτι για τον καθένα από αυτού του τομεί ξεχωριστά. Ευχαριστώ, συνάδελφε Κέλλη. Ολοκληρώσαμε τι επεξηγήσει ψήφου για ε, την 25η επέτειο τη Σύμβαση στο ΙΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Και περνάμε τώρα στι επεξηγήσει ψήφου για τι προτάσει ψηφίσματο ε, για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Ξεκινάει η συνάδελφο Γκίλ. Uh, Ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει τις ε, υποσχέσεις της όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά. Όχι μόνο έχουμε απώλειες 260 ε, εκατομμυρίων ευρώ ε, λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στην ανάκαμψη από την οικονομική κρίση. Η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα μας επιτρέψει να βάλουμε την Ευρώπη στο δρόμο προς την καινοτομία, την δημιουργία θέσεων ε, και την ανάπτυξη. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθήσει να ε, σταματήσει την ε, ανάπτυξη της Google, διότι η αποτελεσματική ενιαία αγορά εξαρτάται από ίσες συνθήκες ανταγωνιστικότητας ώστε να υποφελούνται και οι χρήστες και όλες οι εταιρείε και όχι μόνο μία μεγάλη εταιρεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μπούντα. Πρόεδρε, υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό. Η ενιαία ψηφιακή αγορά σημαίνει εφαρμογή του τρίτου κύματος της τεχνολογικής επανάστασης, της ψηφιακή επανάστασης. Η διασύνδεση των αγορών αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η, η ικανότητα να προσαρμοστούμε στις τεχνολογικές αλλαγές είναι προπόθεση για την ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να το κάνουμε αυτό για να έχουμε ε, καλά αποτελέσματα και νέες θέσεις εργασίας. Η ψηφιακή αγορά ωστόσο, ε, περιέχει πολλές ε, προκλήσεις. Η πολυμορφία των εθνικών αγορών αποτελεί εμπόδιο και υπάρχουν επιτυχείς πρωτοβουλίες όπως είναι η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη για τις ε, δημόσιες ε, συμβάσεις. Επίσης έχουμε τις ε, δραστηριότητες e-commerce οι οποίες έχουν βοηθήσει οι εταιρείες αλλά υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές και διακόπτει ο πρόεδρος τον ομιλητή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα αυτή την ψηφιακή ενιαία αγορά που μας παρουσιάζεται ότι έχει τεράστιες δυνατότητες για να αναζαγωνίσει την ε, ανάπτυξη και ε, την ε, κατανάλωση. Μετά την ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θέλει να επελευθερώσει και την ψηφιακή αγορά. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό στις ψηφιακές νέες αγορές και υπολοιπόμεθα πολύ στην Ευρώπη. Ε, η Ήπεθρο σε μεγάλο βαθμό ας πούμε δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Θα πρέπει όμως να φροντίσουμε να μην είναι δούριο ύπος αυτή η απόπειρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα σαρώσει την εθνική κυριαρχία. Ε, η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και η ελευθερία για όλους τους Ευρωπαίους και τις επιχειρήσεις να έχουν ε, τις ψηφιακές υπηρεσίες που επιθυμούν από όπου και αν προέρχονται για να μην υπάρχει κανένα dumping ε, όπως γίνεται με τα βίντεο on demand και τα Netflix πρέπει να είναι δεδομένη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπίλντε. Ο κύριος Πόσπισιλ. Ευχαριστώ πρόεδρε υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό και το συνυπέγραψα. Να πω απλώς δύο λόγια για τις τελευταίες ε, κουβέντες που μεταφέρθηκαν ε, και μεταδόθηκαν ξανά και ξανά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είμαστε κατά τον Google, δεν κατονομάζουμε κάποια εταιρεία. Απλώς λέμε ότι η Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή θα πρέπει να ε, προβλέψει διαχωρισμό των μηχανημάτων διερεύνησης των ψαχτηρίων από το υπόλοιπο διαδίκτυο των μηχανών αναζήτησης. θα πρέπει να μην επιτρέψουμε να παραμείνουν τα μονοπόλια, τα μονοπόλια που ποτέ δεν ωφελούν τους καταναλωτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξεύρει κάποιες λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σιάρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή για τρεις λόγους τουλάχιστον. Ε, καταρχάς ε, είχαμε καθυστερήσεις ε, όσον αφορά τη σύγχρονη υποδομή του 21ου αιώνα. Έχουμε μια εσωτερική αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κινητικότητα αλλά να αποφύγουμε και τα μονοπόλια. Και όσον αφορά τα δίκτυα και τα κινητά τηλέφωνα, βλέπουμε ότι η τεχνολογία δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Ε, ευτυχώς μπορέσαμε να καταργήσουμε μαζί ε, τις, τα τέλη roaming των εταιριών ε, και άλλα τέτοια κρυμμένα κόστη και είναι σημαντικό το θέμα αυτό και για την Ήπεθρο. Ε, Χρειάζεται λοιπόν η ψηφιακή δικτύωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε Γιάρη, η συνάδελφος Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, διότι χρειαζόμαστε δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού. Ε, τρεις παρατηρήσεις να κάνω. Ε, νωρίτερα είχαμε, τα σημεία, είχαμε σημεία συμφόρησης όσον αφορά την πρόσβαση στο ίντερνετ. Ε, αυτό ε, υπήρχε στους παρόχους υπηρεσιών, αλλά ε, τώρα ε, αυτά υπάρχουν ε, στους στους υπεύθυνους των δικτύων. Δεύτερον, χρειαζόμαστε μια πολιτική συζήτηση σχετικά με το unbundling. Ε, θεωρώ ότι αυτό το μέσο είναι υπερβολικό. Χρειαζόμαστε όμως ε, ίσες συνθήκες εργασίας, γι' αυτό πρέπει να ε, το συζητήσουμε αυτό πολιτικά. Και τέλος, δεν θέλουμε να κατονομάσουμε συγκεκριμένε επιχειρήσεις. Ως βουλευτές νομίζω ότι είναι δίκαιο να εξετάσουμε τι ακριβώς συμβαίνει ε, στον ψηφιακό κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ, ο συνάδελφος Κέλλη. Ευχαριστώ. Φυσικά όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόσουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν αυτή την ενιαία ψηφική αγορά για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την ε, οικονομική ύφεση και να έχουμε ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καταψηφίσαμε όμως ε, την ε, τροπολογία 10, το δεύτερο μέρος, που μιλάει για το unbundling όσον αφορά τις μηχανές αναζήτησης. Και νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για ένα τέτοιο βήμα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε βέβαια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Ιδιαίτερα πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να έχει συνέπειες στη χώρα μου και σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Τελειώσαμε λοιπόν με το θέμα αυτό για την ενιαία ψηφιακή αγορά και ερχόμαστε στον υποσυντισμό των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η κυρία Αγγέλη έχει το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι απαράδεκτο 417 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών να υποσυτίζονται σε χώρες με ανάπτυξη και 5 εκατομμύρια παιδιά να έχουν σοβαρό υποσυτισμό. Θα πρέπει αυτοί οι αριθμοί να λειτουργήσουν ως σήμα συναγερμού για μας. Όχι μόνο για να εντείνουμε τον, ε, την ε, τον συντονισμό των πολιτικών ανάπτυξη και επισητισμού, αλλά να δούμε ότι υπάρχει αυτό ο απαράδεκτος ε, πόνο ε, σε αυτέ τι περιπτώσει λόγω πολιτική ανεπάρκειας, όχι μόνο των πολιτικών, ε, των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτέ τι χώρε εμεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε, δίνοντα τι προσπάθειές μα για να βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτό το ζωτικό τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χαραντέν εδώ. Ο κύριος Μοργκάνο; Μοργκάνο. Ευχαριστώ πρώτα Την περασμένη εβδομάδα η Διεθνή Διάσκεψη για τον Εξωτισμό τη ΦΑΟ έδωσε αριθμού εντυπωσιακού. 850 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο έχουν ε, χρόνιο υποσυτισμό. 160 εκατομμύρια παιδιά ε, σε χώρε με καθυστέρηση υποσυτίζονται. 5% το ε, των 9 εκατομμυρίων θανάτων παγκοσμίω οφείλονται σε υποσυτισμό. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντείνει τη δράση τη σε διεθνέ επίπεδο, να κοινοτοποιηθεί και να εξεύρει κονδύλια και πόρου μακροπρόθεσμου ε, σε συνεργασία με του φορεί του ΟΗΕ, του G8 και του G20, με του άλλου ε, παγκόσμιου οργανισμού και με μη κυβερνητικέ οργανώσει, ώστε τα κράτη, μεταξύ των οποίων και αυτά τη ΕΚΠΟ 2015, να αναλάβουν δεσμευτικού στόχου στόχους για την καταπολέμηση της ένδυας και του υποσυτισμού με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εντατική μεταξύ του συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Με Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Ε, το θέμα αυτό συνδέεται και με το προηγούμενο για την 25η επέτειο ε, της Σύμβασης του ΙΟΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Βέβαια, το πρώτο που χρειάζεται ο άνθρωπος στη ζωή του είναι να έχει αρκετό φαγητό ε, και ε, αρκετή ποικιλία. Αυτό δεν συμβαίνει παντού στον κόσμο και δυστυχώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αξίζει να δέχεται επικρίσεις γιατί οι επιδόσεις μας είναι γνωστές. Είμαστε υπαριθμόν ένα στην ανθρωπιστική βοήθεια. Βέβαια πάντα χωράει βελτίωση και τα θέματα που αναφέρει το ψήφισμα χρειάζονται προσοχή για να δούμε πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Ιδιαίτερα να βοηθήσουμε τις χώρες να αντιμετωπίσουν, να έχουν καλύτερη ε, και πιο αηφόρο γεωργία, πούμε, και γενικότερες πρακτικές. Ε, χάρηκα ε, για το ψήφισμα αυτό και με χαρά το υποστήριξα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ταραμπελά θα βάλει την κοινοβουλευτική τελεία αυτή τη βδομάδα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα για τον υποσυτισμό των παιδιών ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Καλύτερα θα ήταν, έχει ε, γίνει δεκτή και η τροπολογία 3, γιατί ε, ο, και ο Λιβιέντε Χιούτερ, ειδικό ηγητής του ΟΗΕ, αυτά λέει στην έκθεσή του για τις προτεραιότητες στην αναπτυξιακή πολιτική της Γεωργίας, αλλά ε, το ΕΛΚ που μας κοπανάει συνέχεια αυτά που είπε εδώ ο Πάπας να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και την ανισότητα αλλά δεν κατάλαβε το μήνυμα ο Πάπας Φραγκίσκος δεν θα πρέπει να είναι πολύ περήφανος για τους πιστούς τους εδώ που την ώρα του μηνύματος χειροκροτούν αλλά δεν μεταφράζουν τα χειροκροτήματα σε ψήφο και γινούν την πλάτη στις βασικές αρχές που είναι τόσο απαραίτητες για τη μέση της φτώχειας Ευχαριστώ κύριε Ταραμπέλα Τελειώνουν εδώ οι επεξηγήσεις ψήφου για το ψήφισμα αυτό υποσυντισμό στο πεδίο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ορίστε. Κύριε Κέλλη, διαδικαστικό βάζετε. Ναι, ένα διαδικαστικό. Ήθελα να το πω και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, αλλά δεν θέλησα να καθυστερήσω το σώμα, ούτε και εσάς να σας φέρω σε δύσκολη θέση, Πρόεδρε, γιατί είστε υποδειγματικός στην Προεδρία σας. Έχει να κάνει με την προφορική τροπολογία αν δεν ήταν η 11 σε σχέση με τη μελέτη αντικτύπου. Έγινε ε, ονομαστική κλίση και μετά ο εκπρόσωπος των φιλελευθέρων σηκώθηκε και έκανε προφορική τροπολογία. Τουλάχιστον εγώ έτσι το κατάλαβα. Κανονικά η προφορική τροπολογία παρουσιάζεται πριν να τεθεί σε ψηφοφορία η ε, εν λόγω παράγραφος. Αυτό ήταν δηλαδή τροπολογία ή επεξήγηση ψήφου. Αυτό θέλω να διευκρινιστεί. Έχω και την απάντηση. Αλλά... Κύριε Κέλλη, ε, θελήσατε να έχετε εσείς τον τελευταίο <laughs> λόγο. Δεν σας άρεσε αυτό που είπα ότι θα βάλει τελεία ο κύριος Ταραμπέλα. Ε, ψηφίσαμε την τροπολογία 11 ονομαστικά και μετά σηκώθηκε ο συνάδελφος που δεν θυμάμαι τώρα ε, από τους φιλελευθέρους και έκανε προφορική ε, τροπολογία στην παράγραφο 11, στο αρχικό, όχι στην τροπολογία 11, στην παράγραφο 11. Ήταν σε άλλο σημείο στην ε, λίστα ψηφοφορίας και αυτή η προφορική τροπολογία εγκρίθηκε. Ωραία. Τα πρακτικά θα διανεμηθούν στην επόμενη σύνοδο και αν δεν διαφωνεί κανείς θα θεωρήσω εγκεκριμένα τα ψηφίσματα. Μάλλον θα τα διαβιβάσω αρμοδίως τα όσα εγκρίναμε. Ευχαριστώ πολύ που παραμείνατε πέντε συνάδελφοι. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες και ιδίως τους διερμηνείς στις καμπίνες